Τα πρακτικά της συνεδρινής συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στην αρχή της επόμενης συνόδου. Και τότε θα εγκριθούν και θα σταλούν στους δικαιούχους. Λίγη εδώ προσωρινά διακόπτεται η σύνοδος και... Σας εύχομαι καλή επιστροφή. Ευχαριστούμε.